ήσασταν ο τελευταίο ομιλητής ε, για επεξήγηση ψήφου, θα σας κάνω μια ανακοίνωση. Πήραμε από το Συμβούλιο ε, θέση του Συμβουλίου και του, ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μια κοινή θέση. Μπαίνω στο πειρασμό να σας διαβάσω το τίτλο. Είναι μια κοινή θέση της 5ης Μαρτίου του 2009 εν ώψη έγκρισης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενός κανονισμού που ε, αφορά τις, ε, ε, τους, διπλωμάτες ε, σταδιοδρομίας ε, σε σχέση με την υποβολή και αποδοχή των αιτήσεων θεώρησης. Για να σας δείξω ότι τα πράγματα είναι πολύπλοκα καμιά φορά στην Ευρώπη από αύριο, 13 Μαρτίου, ε, έχουμε ε, αρχίσει η η διαδικασία ε, που θα διαρκέσει τρεις μήνες για την υποβολή τροπολογιών. Κύριε, ε, ο κύριος Ανάν λέει, παραλείψατε να μου αναφέρετε το όνομά μου για το Θιβέτ. Έχετε το λόγο. Οι Θιβετιανοί, κύριε Πρόεδρε, όπως όλα τα έθνη, έχουν το δικαίωμα να ζουν βάσει των δικών τους ε, κανόνων και αρχών. Αρνούμενοι το δικαίωμα τους αυτό, ε, είναι, σημαίνει ότι λέμε ότι οι Σοβιετιανοί δεν καταλαβαίνουν ποιο είναι το θέμα. Ε, δεν έχουν δικαίωμα στη δημοκρατία. Κάνω μια έκκληση προς το Κοινοβουλίο να ε, δει την ηρωνία στη σχέση Ανάμεσα σε αυτά τα επιχειρήματα και αυτά που ακούστηκαν μετά το όχι στα δημοψηφίσματα τη Ολλανδία, τη Γαλλία και τη Ιρλανδία. Ότι δηλαδή δεν ε, καταλάβαιναν ε, ποιο ήταν το θέμα. Ότι ψήφιζαν κατά του Ιράκ, κατά τη Τουρκία, κατά του αγγλοσαξονικού φιλελευθερισμού κλπ. Και ότι χρειάζονταν καλύτερη ενημέρωση. Εγώ πιστεύω ότι είτε μιλάμε για το Θιβέτ, είτε για τα κράτη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ο λαό κατανοεί πάρα πολύ καλά τι επιθυμίε του ε, και θα πρέπει να είναι ελεύθερο να ε, εκφράζει τις επιθυμίες του αυτές με την ψήφο του. Και γι' αυτό ε, επαναλαμβάνω ότι θα πρέπει να ε, ξανακάνουμε το δημοψήφισμα για τη συνθήκη της Λισαβόνας. Ευχαριστώ. Θα διακοπεί εδώ η συζήτηση, λέει ο Πρόεδρος. Θα επανέλθουμε στη θέση ώρα για να ζητήσουμε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη δημοκρατία και του κράτου δικαίου. Έχουμε Γουινέα Μπισάου, Φιλιππίνε και Νταρφούρ. Ε, διακόπτουμε εδώ. Σα εύχομαι καλή όρεξη.